Αγαπητοί συναδελφοί, θα ολοκληρώσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου και προχωρούμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Κλάς. Η κυρία το βαγιά, ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,